το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και προσβλέπω σε αυτήν τη συνεργασία με όλους σας για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ πολύ.